Good morning. Uh, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και όλους. Καλωσορίσατε στη συνεδρία της Επιτροπής Προπολογισμών. Το πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης είναι η έγκριση αυτής. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θεωρώ ότι εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη και περνούμε στο δεύτερο σημείο. Ανακοινώσεις ε, του Προέδρου Δύο έχω να σας ε, μεταφέρω. Πρώτον, αποφάσεις συντονιστών της 23ης Ιουλίου. Είναι στο φάκελό σας το σχετικό έγγραφο και αν δεν έχετε αντιρρήσεις θα θεωρήσουμε ότι εγκρίνεται το έγγραφο αυτό. Δεύτερο, πριν τι θερινέ διακοπέ, κάλεσα τη Φινλανδική Προεδρία να έρθει να παρουσιάσει το πρόγραμμά της και τις προτεραιότητές της στα μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Πρόκειται για μια καθιερωμένη πρακτική. Οι υπουργοί δηλαδή της κάθε εκπεριτροπής προεδρίας... Παρακαλώ, αν μπορώ να έχω λίγη ησυχία. Έλεγα λοιπόν ότι είναι καθιερωμένη πρακτική να έρχονται οι υπουργοί της εκάστοτε εκπεριτροπή Προεδρίας στις Επιτροπές και να ε, συζητούν για τα ε, προγράμματα και για τους ε, Βέβαια, το Συμβούλιο ε, δεν έρχεται ε, συχνά εδώ, παρότι σε άλλες επιτροπές πηγαίνει. Έχω σταμένος μιλήσει για την διοργανική συνεργασία. Ε, Παρ' όλα αυτά και η Φιλανδική Προεδρία απέρριψε την πρότασή μου και το θεωρώ αυτό άκρο λυπηρό, ιδίω από τη στιγμή που τώρα ε, θα επαναλάβουμε τι εργασίε μα για πολύ σημαντικά ζητήματα, όχι μόνο το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, αλλά και έχουμε στρατηγικού φακέλου σε θέματα συναπόφαση, ε, rule of law, πρόγραμμα στήριξη μεταρρυθμίσεων και λειτουργία σταθεροποίηση στι. 4 Σεπτεμβρίου θα υπάρξει ανταλλαγή απόψεων των Υπουργών με τα μέλη τη Επιτροπή ΕΚΟΝ για ζητήματα που είναι και κοινή αρμοδιότητα ΕΚΟΝ Badge. Μιλάω δηλαδή για αύριο. Θα ήθελα να συμμετάσχετε όσοι μπορείτε στη συνδρίαση αυτή, γιατί φαίνεται να είναι η μόνη δυνατότητα να μπορέσουμε ως Επιτροπή Προπολογισμού να συζητήσουμε το Συμβούλιο τα θέματα που είναι δικέ τη αρμοδιότητα. Ελπίζω βέβαια να, θεωρεί στο μέλλον αυτή την προσέγγιση το Συμβούλιο, διότι δεν μπορεί να δικαιολογηθεί και δίνει και ένα πολύ λάθος μήνυμα. Αντί δηλαδή να συνεργαζόμαστε, ε, γίνεται το αντίθετο. Αυτά σε ό,τι αφορά τι ανακοινώσει μου. Τρίτο σημείο, έγκριση πρακτικών. Αντιρρήσεις αν όχι εγκρίνονται. Και τώρα περνάμε στην ώρα ψηφοφορίας. Καλό θα τα κάνουμε πρώτα μία δοκιμή. Εντάξει. Α, πρέπει να βάλουμε τις κάρτες όμως πρώτα στο μηχάνημα. Ψηφίζουμε. Τι πρέπει να κάνουμε. Μάλιστα, πρέπει να ψηφίσουμε. Πιέστε να κουμπί εκεί κάποιο, τέλος πάντων. Πέρας ψηφοφορίας more than allowed. So one renew member should not vote. Okay, the electronic. Ε, ένας από τη Renew είναι υπεράριθμος από ό,τι μου λέει εδώ ο ειδικό. One, one renew vote too much, I'm sorry to say. It's okay? Το ρυθμίσαμε. Ωραία, άρα λειτουργεί το σύστημα, από ό,τι φαίνεται. Σημείο 4. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθμών 1. Για το Γενικό Προπολογισμό του 2019 προτείνω να ψηφίσουμε την τροπολογία διανατάσσεως χειρός ψήφι υπέρ. Στροπολογίας 1. Όχι, δεν ψηφίζουμε με τις, κάρ, με κάρτες μας, ψηφίζουμε αναδιανατάσεως. Ψήφι υπέρ της τροπολογίας 1. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται λοιπόν η τροπολογία. Και προχωρούμε στην τελική ψηφοφορία του σχεδίου εκθέσεως, όπως δεν τροποποιήθηκε, λέει ο πρόεδρος. Ονομαστικά θα ψηφίσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας 37 είναι ψηφίσαντες, 32 ψήφοι υπέρ, 4 κατά και μία αποχή. Συγχαίρω τον Τζον Χάουερ. Πού είναι? Α, εκεί, μάλιστα. Συγχαρητήρια λοιπόν για αυτήν την έκθεση και σας ευχαριστώ. Προχωρούμε στο σημείο 5, το σχέδιο διορθωτικού προεπλασμού παριθμών 2 να ψηφίσουμε καταρχάς τροπολογία Σαστέλ. δυνατά στις χειρός ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Α, η τροπολογία γίνεται δεκτή. Ηλεκτρονικά τώρα ψηφίζουμε το σχέδιο έκθεσης. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε ψηφοφορία 39, οι ψηφίσαντες 31 ψήφοι υπέρ, 7 κατά, μία αποχή. Που σημαίνει ότι το σχέδιο έκθεση όπως τροποποιήθηκε γίνεται δεκτό. Και συγχαίρω τον εισηγητή που είναι για μια ακόμη φορά ο κύριος Χάρτ. Περνάμε στο σημείο 6. Πρόταση απόφασης ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς τη Ρουμανία, την Ιταλία και την Αυστρία. Δεν υπάρχουν τροπολογίες, άρα προχωρούμε απευθεία στην ηλεκτρονική ψηφοφορία που του σημείου αυτού, του σημείου 6, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 35 ψήφοι υπέρ, μία κατά, τρεις αποχές. Άρα γίνεται δεκτή. η έκθεση στο σημείο 6 και συγχαρητήρια στον κύριο Μουρέσα. Περνάμε στο 7. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού παριθμών 3 σχετίζεται με την απόφαση που μόλις λάβαμε ε, πριν, το 6 δηλαδή, Πρόκειται πάλι για την πρόταση κινητοποίηση του Αμεριλεγγύη Ευρωπαϊκή Ένωση για την παροχή βοήθεια στι τρει χώρε που προανέφερα. Δεν έχουμε κάποια τροπολογία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Περιμένω τρεις ακόμη συναδέλφους ε, και τώρα κλείνει λίγη ψηφοφορία. 36 ψήφοι υπέρ, καμία ψήφο κατά, τρεις απόχέ. άρα εγκρίνεται και αυτό το σχέδιο διορθωτικού προβλησμού και αυτή η έκθεση συγχαίρω τον Τζον Χάουερθ. Σημείο 8 Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής. Έχουμε τέσσερι τροπολογίες. Θα ψηφίσουμε διατάσσως της χειρός την τροπολογία 3 καταρχάς, ψήφι Κατά. Αποχές. δεκτή. Τροπολογία 4. Ψήφι περ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Ψήφι Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Ψήφι περ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και τώρα έχουμε τις αιτιολογικές σκέψεις. Ε, recital 1. Ψήφι περ κατά αποχές εγκρίνεται. Και σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες τροπολογίες, τροπολογίδι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Οι και προχωρούμε στην τελική ψηφοφορία της έκθεσης όπω τροποποιήθηκε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. 31 ψήφοι υπέρ, 3 κατά, 5 αποχές είναι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Συγχαρητήρια στον κύριο Ρόντσα. Σημείο 9. Επιτροπή. Δεν υπάρχει κάποια αίτηση μεταφοράς, άρα περνάμε κατευθείαν στο σημείο 10, μεταφορές ε, σε άλλα τμήματα και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Φερνάντες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δύο αιτήσει μεταφοράς έχω. Για τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή για τη μεταρρύθμιση διαφόρων γραμμών 1612 επίσης 15.000 ευρώ για νομικά ζητήματα και άλλα. 2.000 ε, για ενίκεια, 22.000 ε, για το Μοντουαγέ στην Ρίσιντες εδώ στις Βρυξέλλες. Επίσης, δυνάμει του 231 έχουμε 85 περίπου χιλιάδες ε, παραπάνω χρήματα για την ε, υπηρεσία μετάφρασης ε, και στην 3400 στα διάφορα και μια τρίτη μεταφορά που καλύπτεται εδώ. Είμαστε υπέρ, άρα εμείς ε, εγκρίνουμε και τα τρία αυτά αιτήματα και το C8 2019 σας παρουσιάσω τώρα. Ο στόχος είναι ε, να τηρηθούν οι διατάξεις ε, του μισθολογικού καθεστώτος ε, των βουλευτών και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι δεν εξελέγησαν το 5% των βουλευτών, των απερχόμενων όπως προ, είχαμε προβλέψει, αλλά λιγότεροι. Και Έχουμε λοιπόν γύρω στα 3,5 εκατομμύρια πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και και τη γραμμή 1006. Μεταφορά για να αντιμετωπιστούν κάποιες νομικές υποχρεώσεις ε, όπως αυτές προκύπτουν από το καθεστώς των βουλευτών και για την συγκεκριμένη μεταφορά C8 λοιπόν ζητώ να ψηφίσετε υπέρ για τον προϋπολογισμό ε, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για τον διαμεσολαβητή. 4. 2019. Ναι, υπήρχε μια μικρή καθυστέρηση, λέει ο πρόεδρος, αλλά τέλος πάντων. Ε, οι σκιώδεις εισηγητές θα ήθελαν μήπως το λόγο. Η κυρία Γκαρτιά Θάμπαλ, κάποιος άλλος. Υπάρχει κάποιος οποιοδήποτε που θέλει το λόγο, όχι. Άρα, να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, όχι για το διαμεσολαβητή. αλλά για τα άλλα ζητήματα που έχουμε. Αν δεν υπάρχει αντίρρηση σε σχέση με το διαμεσολαβητή, εγώ θα έλεγα να μην ψηφίσουμε. Βέβαια, αν εσείς θεωρείτε ότι χρειάζεται να ψηφίσουμε. Αλλιώς όχι, ψηφίζουμε το άλλο θέμα. The Κυρίσω την έναρξη της ψηφοφορίας. I declare the vote closed. We have 28 in favor. 28 υπέρ, 7 κατά, μία αποχή. So, adopted. Εγκρίνεται. Και συγχαρητήρια στον κύριο Φερνάντες. Policy. I'd like to give the πολιτική κτηρίων. Και έχουμε τον πάγιο μόνιμο εισηγητή μας, την κυρία Κέλλερ. Ευχαριστώ. Όπως και εσείς και εγώ να καλωσορίσω τους ε, συναδέλφους με τις διακοπές αλλά και τους διερμηνείς μας. Όσον αφορά τώρα αυτό το σχέδιο κειμένου Έχουμε την ε, ανοικοδόμηση νέων γραφείων. Αφορά την ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Το 2017 ξεκίνησε αυτή η υπόθεση και ήδη έχει υπάρξει έγκριση από το Κοινοβούλιο τον Ιανουάριο του 2018. Σας υπενθυμίζω ότι έχουν εγκαταλειφθεί τα γραφεία που είχαμε γιατί που ήταν πολύ ε, απαρχαιωμένο. Και επίσης είχαμε και λήξη κάποιων μισθώσεων. Οπότε έγινε κάποιος διαγωνισμός από την υπηρεσία εξωτερικής δράσης και επελέγει μια συγκεκριμένη πρόταση. Αυτό αφορά και κάποια ε, επιχείρηση που θα βοηθήσει να ε, εκτελέσει τις εργασίες, να βρει και τον το μέρος που θα κατασκευαστούν αυτά τα γραφεία και δημιουργικά αυτό συζητούμε σήμερα, Ζητείτε μια αύξηση της αρχικής προοικοδότησης για 5,4 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε το ετήσιο μίσθωμα από 4,5 πάει στα 5,1 εκατομμύρια για το σύνολο της μισθώσεως έχουμε 98,8 εκατομμύρια ευρώ αντί για 93,3. Συγγνώμη για όλα αυτά τα νούμερα. Αλλά πάντως σας ε, ζητώ να εγκρίνετε την πρόταση για αυτές τις εργασίες γιατί είναι θέμα ασφαλείας με θωρακισμένες πόρτες, ε, με ανοιχνευτές μετάλλων, σκάνερ και από το 2018 μέχρι σήμερα με έκπληξή μου είδα ότι χρειάζεται να υπάρξουν συμπληρωματικές εργασίες παρά το ότι υπάρχει επαρκής ε, πρόβλεψη ασφαλείας. Όμως αυτό είπαν οι αρμόδιες ε, υπηρεσίες και γι' αυτό δεν είχαν ε, ληφθεί υπόψη αυτά τα στοιχεία στην αρχική πρόταση που είναι από μισή χρόνο. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Εμείς ευχαριστούμε κυρία Κέλλερ. Δύο παρατηρήσεις. Έχουμε την ομαδεργασία του Συμβουλίου που μελετά αυτή την πρόταση σήμερα κιόλα. Δεύτερον, οι, οι εκπρόσωποι ε, της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης παρίστανται και ε, Ήδη σας έχει υποβληθεί κύριε, ε, μια ερώτηση από την κυρία Κέλλερ, οπότε μπορεί να λέτε το λόγο για να απαντήσετε αυτή την ερώτηση της κυρίας Κέλλερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε για την παρουσίαση του φακέλου. Δεν θα καθυστερήσω και θα απαντήσω στην ερώτησή σας γιατί είναι σημαντικό να γίνει σαφές λίγο πιο δυνατά παρακαλώ να πλησιάσω το μικρόφωνο ακούγομαι καλύτερα μάλιστα έλεγα ότι είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη ότι δεν συζητούμε για κάποια συνήθεια κτίρια γραφείων. Ο σκοπός αυτών των νέων γραφείων είναι να αντικατασταθούν τα δύο κτίρια της λεωφόρου Κόρτεμπεργκ. όπου τώρα στεγάζεται το στρατιωτικό προσωπικό. Οι προδιαγραφές ασφαλείας για αυτές τις υπηρεσίες πρέπει να είναι πολύ πάνω από τον μέσο όρο για τα συνήθη γραφεία, τα συνήθη κτίρια τέτοιων υπηρεσιών. Δεν πρόκειται μόνο για το προσωπικό. Είναι και θέμα διαφόρων διαβαθμισμένων πληροφοριών, ε, περιορισμένη πρόσβαση σε κάθε γραφείο, ασφαλής επικοινωνίας. σε υψηλό επίπεδο ε, διαβάθμισης και γι' αυτό και τα στάνταρ είναι πολύ παραπάνω από τα συνήθεια. Εξού και το υψηλότερο αντίστοιχο κόστος. Έτσι εξηγείται λοιπόν αυτό το παραπάνω κόστος. Τώρα, γιατί σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα ε, έτσι έγινε και άλλαξε η, η Οπότε, η ανακαίνιση ξεκίνησε σχεδόν ταυτόχρονα όταν ε, διατυπώθηκε το ποιες είναι οι απαιτήσεις ασφαλείας. και αυτά όλα τα είχαμε εισηγηθεί στην αρχή επί του προϋπολογισμού τότε και είχαμε επισημάνει ότι υπήρχε ένα περιθώριο το οποίο θα έπρεπε να εξειδικευτεί αργότερα γιατί αυτές οι προοδευτές ασφαλείας θα έπρεπε και αυτές να συγκεκριμενοποιηθούν στη λεπτομεριά τους. Έγινε αυτό. Οπότε γι' αυτό και σήμερα βρισκόμαστε εδώ ακριβώς γιατί ανέβηκε ο πύχης περισσότερο. Έτσι, παρεμπιπτόντως να σας πω ότι για να υπάρχει πρόσβαση ε, μέσω δακτυλικού αποδεικτυπώματος σε κάθε γραφείο συνεπάγεται ένα κόστος. Μια που χρειάζονται σε κάθε όροφο του κτηρίου 11 χιλιόμετρα καλωδίων. Αυτό έτσι σαν πει κάτι και λεπτομέρειες σας το λέω ε, για να καταλάβετε τι σημαίνει όλο αυτό το έργο. Ήδη υπάρχουν αυτά τα καλώδια και Εάν είχαμε το σύνθεσ ε, επίπεδο ασφαλείας, τότε όλα αυτά θα ήταν μια τρύπα στο νερό, θα ήταν ε, μια διασπάθηση του κοινωτικού χρήματος. Οπότε, παρά την ευξημένη δαπάνη, παραμένει το κτίριο να έχει κάποιο ενδιαφέρον ως πρόταση. Ό,τι άλλο θέλετε, ευχαριστώ να σας το εξηγήσω. Ευχαριστώ, λέει Θέλετε να απαντήσετε κυρία Γέλερ. Όχι. Έχετε άλλε ερωτήσεις ή παρατηρήσεις μια που φιλοξενούμε τους εκπροσώπους της υπηρεσία εξωτερικής δράση Ωραία. Τότε ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε. Το κείμενο τη συγγήτριας ψηφίζουμε. And closed. Πέρασε. with a result of 28 in... 28, 7, με δύο εποχές. Συγχαρητήρια, κυρία Κέλλερ. Time is uh, over. Έτσι ολοκληρώθηκε ε, κομμάτι της ψηφοφορία και πάμε τώρα στο σημείο 12 της ε, πρωινής συνεδρίασης που αφορά τον Γενικό Προεδρικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την χρήση του 2020. Οπότε θα με την σκητάλη στην ε, Γενική Σύγκριτη, την κυρία Μόνικα Χολμαϊρ, Καλημέρα σας κυρία. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα παρουσιάσω το περιεχόμενο ενός εγγράφου εργασίας σήμερα μετά τον πρώτο τριμερή, ας πούμε, διάλογο, το ολοκληρώσαμε. Ε, βέβαια ήταν λίγο απογοητευτικό το αποτέλεσμα γιατί το Συμβούλιο δεν έδειξε καν την προθυμία να κάνει σοβαρό διάλογο και στο τέλος ο Πρόεδρος έκανε πολύ εύστοχες παρατηρήσεις ε, αφού όταν, όταν, όταν, ε, όταν κάποιος ε, λέει ότι θα κάνει αντικειμενικές περικοπές πρέπει να είναι αντικειμενικές και τα επιχειρήματα αντικειμενικά όχι να διευρύνουμε το περιθώριο χωρίς αντικειμενική ε, αιτιολόγηση. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάντως ως εισηγήτρια τους ε, σκιώδεις και τους συντονιστές για την υποστήριξη. Ευχαριστώ και για την υποστήριξη της Γραμματείας, για τη σύνταξη του εγγράφου εργασίας και για την προθυμία να διαθέσει όλα τα στοιχεία και έγγραφα για να γνωρίζουν καλά όλοι οι συνάδελφοι πού βρίσκονται τα προβλήματα και όλα αυτά μπορεί κανείς να τα δει αν θέλει και λεπτομερώς. και τα βασικά στοιχεία θα τα γνωρίζουν. Λοιπόν, ποια είναι τα βασικά θέματα για τις περικοπές. Το Συμβούλιο τι θέλει να περικόψει. Το Συμβούλιο στο, ε, στην επιστήμη και έρευνα βάζει το θέμα της ψηφιοποίησης, βάζει και θέματα κλίματος, ε, και τις μικρομεσαίες. Αυτό ε, δείχνει ότι λείπει μια βασική γνώση και κατανόηση. Η Φιλανδική Προεδρία τι είπε. Θέλει περισσότερη ψηφιοποίηση, περισσότερη καινοτομία, περισσότερη τεχνολογική ανάπτυξη ε, μέσα στα πλαίσια του προγράμματος πλαισίου ε, το Συμβούλιο ε, είναι εκ διαμέτρου αντίθετο με την Φιλανδική Προεδρία. Ε, στον τομέα της έρευνας και της, ανα... της επιστήμης, το μεγαλύτερο κομμάτι των περικοπών πλήττει τα θέματα αυτά. 15% του προϋπολογισμού είναι αυτό. Οι περικοπές όμως είναι το 50% των προτινομένων περικοπών από το Συμβούλιο σε ένα πρόγραμμα που είναι 15% του προϋπολογισμού. Είναι λοιπόν δύσκολη αυτή η διαδικασία που ακολουθεί το Συμβούλιο και δεν υποστηρίζεται επαρκώς, δεν επαληθεύεται. Επίσης, το Συμβούλιο απορρίπτει το 15.3 του Δημοσιονομικού Κανονισμού, διότι αυτό το άρθρο θα ισχύει μόνο σε ειδικέ περιπτώσεις. Το 15.3 άρθρο του Δημοσιονομικού Κανονισμού αναφέρεται συγκεκριμένα όμως στην επιστήμη και την έρευνα. Όχι σε μέσα αντιμετώπιση της κρίτησης, δεν είναι ταμείο αλληλεγγύης ή παγκοσμιοποίησης, είναι για να ενισχύει την έρευνα, την επιστήμη και μόνο για αυτό το τομέα προβλέπεται. Όταν λοιπόν ε, εντοπίζει κανείς κάποιο έλλειμμα, κάποιο πρόβλημα στην επιστήμη και την έρευνα, τότε στα προγράμματα ε, που είχαμε προβλέψει κυρίως ως κοινοβούλιο, βασικά, ε, όταν υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη, πού βρίσκεται ιδιαίτερη ανάγκη σε όλα τα προγράμματα που έχουν πολύ μικρό ποσοστό επιτυχίας. Τι σημαίνει το ποσοστό επιτυχίας. Έχουμε 100% των προτάσεων που αξίζει να προωθηθούν, επιλέγουμε τα καλύτερα και να δούμε πόσα θα προωθηθούν και θα χρηματοδοτηθούν. Υπάρχουν προγράμματα που έχουν 90% ποσοστό απόρριψης, όχι γιατί είναι κακά, αλλά γιατί δεν υπάρχουν λεφτά. Γι' αυτά, λοιπόν, θέλαμε πρόσθετη υποστήριξη οικονομική χρηματοδοτική. Και είχαμε μιλήσει και για την αλλαγή του κλίματος στο Σκηνοβούλιο και το θέμα της αναπτυξιακής βοήθειας και στους δύο τομείς ε, υπάρχουν, προτείνονται περικοπές, αλλά και στον τομέα της ψηφιοποίησης γίνεται, προβλέπεται περικοπή. Ε, θα μιλήσουμε και με το Συμβούλιο και με τους Υπουργούς Οικονομικών και με τους ε, ε, πρέσβεις. Εκεί πάντως ε, σημειώνονται οι μεγαλύτερες περικοπές. Εκεί που δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου περικοπές είναι στον τομέα 1β. Στον τομέα 1β υποτομέας 1β. Εδώ ε, υπάρχει η πρωτοβουλία απασχόλησης για τους νέους, η οποία προωθείται ιδιαίτερα. Εδώ δηλαδή ε, αναλαμβάνουν δέσμευση, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί το Συμβούλιο και εδώ κάνει περικοπές, ενώ ουσιαστικά είχαν ανακοινώσει αύξηση. Γιατί δηλαδή ειδικά εδώ πρέπει να γίνονται περικοπές, διότι αυτό αντιφάσκει και στις προτεραιότητες του ε, Συμβουλίου. Ε, επίσης, ε, ε, οι περικοπές των κονδυλίων επικεντρώνονται σε δύο τομείς οποροκυπευτικά και στις αποσυνδεδεμένες άμεσες πληρωμές από το, το Ταμείο Εγγύησης για τη Γεωργία. Πρόκειται για το μίσ που προβλέπεται νομοθετικά η χρηματοδότηση. Αν υπάρξουν περισσότερες αιτήσει πρέπει να πληρώσουμε. Δεν έχουμε άλλη εναλλακτική. Για τα οποροκυπευτικά θα μιλήσουμε πάλι με την, τους συναδέλφους από την Ειδική Επιτροπή για να δούμε αν αυτά όλα είναι θεμητά ε, γιατί έχουμε και το πρόγραμμα για τα φρούτα στα σχολεία και δεν ξέρω αν θέλουμε να κάνουμε περικοπή. Θα δούμε τι θα πούν και οι συνάδελφοι από την Επιτροπή Άγκρη. Στην, ε, στο τομέα 3, ε, εδώ 126,3 είναι οι περικοπές των πιστώσεων υποχρεώσεων, ενώ των πληρωμών είναι κατά 34,5. Όλες οι ε, περικοπές αφορούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες, την Frontex για παράδειγμα μείον 6,6 εκατομμύρια. Θα πρέπει να δούμε αν όλα αυτά είναι δικαιολογημένα. Πρέπει να μιλήσουμε και με τους εκπροσώπους των υπηρεσιών. Το ΆΜΙΦ έχει τη μεγαλύτερη περικοπή. Δεν ξέρω αν έχουμε υποχρέωση ε, να πληρώσουμε χρήματα από το ΆΜΙΦ επιπρόσθετα. Το πρόβλημα της Ελλάδας ε, το βλέπω πάλι να αναβαθμίζεται με την αύξηση των προσφύγων. Μπορώ να φανταστώ ότι η Ελλάδα θα στείλει αιτήματα στην Κομισιόν να πάρει κονδύλια από το ΆΜΙΦ για να προβλέψει καλύτερα ε, για την υποδοχή και διαβίωση των προσφύγων. Θα το δούμε. Στο εσωτερικής ασφάλειας, μείον 25,4 τρόφιμα ζωοτροφές μείον 10 εκατομμύρια. Για το Creative Europe, Δημιουργική Ευρώπη, αυτό πάλι ακατανόητο. Ένα από τα καλύτερα προγράμματα είναι αυτό. Και υποχρηματοδοτείται και μειώνουν και κατά 6,2 εκατομμύριο. Ενώ υποχρηματοδοτείται συνολικά το πρόγραμμα. Τώρα για τα δικαιώματα, την ισότητα, την ηθαγένεια, μείον 2 εκατομμύρια προβλέπετε. Τέλος, μισό λεπτάκι. Τώρα, μοιάζουν οι περικοπές όπως και των προηγουμένων ετών, όμως θέλω να ρωτήσω για το ΆΜΙΦ και το ESF την Κομισιόν αν όντως χρειάζονται λιγότερα κονδύλια ή αν πρόκειται για οριζόντιες επιτρο... Ε, περικοπές. Διότι αλλιώς θα κληθούμε κάποια στιγμή να κάνουμε μεταφορές γιατί θα χρειαστούν χρήματα και θα πρέπει να βρεθούν. Ε, πάντως να το, ρωτούμε, να, το, ρωτήσουμε αυτό, αν δικαιολογούνται αυτές οι περικοπές. Τώρα για το τομέα 4. Εδώ στις υποχρεώσεις ε, ε, Πιστώσει υποχρεών μείων σε 40 εκατομμύρια πρόκειται για το ε, μέσον για την αναπτυξιακή συνεργασία, για την ε, Τουρκία, το, τα προγράμματα, αναπτυξιακή συνεργασία, ανθρωπιστική βοήθεια, ε, το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το Μέσο για την Εταιρική Σχέση και την Ευρωπαϊκή Γειτονία. Εμείς και εδώ θεωρώ ότι θα χρειαστούμε περισσότερα χρήματα από ό,τι λιγότερα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ρωτήσουμε πάρα πολύ συγκεκριμένα ε, αν έχοντας δει όλα αυτά για την υλοποίηση, αν εντωμεταξύ η υλοποίηση προχωρεί 100% και τα προγράμματα αξιοποιούνται πραγματικά. Δεν έχω την εντύπωση ότι χρειαζόμαστε λιγότερα κονδύλια για την αναπτυξιακή βοήθεια. Αντίθετα, για την Βόρεια Αφρική τις χώρες με τις οποίες ε, έχουμε ε, συμφωνία για υποστήριξη και των προσφύγων να αντιμετωπίζονται καλύτερα ε, για τα παιδιά επίσης και τα σχολεία τους, για την σωστή διατροφή. Για όλα αυτά δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα χρειαστούμε λιγότερα κονδύλια και ότι είναι θεμητό να προτείνουμε περικοπή. Ε, τώρα για το προενταξιακό μέσο για την Τουρκία τα προηγούμενα χρόνια είχαμε πει ότι όλη η υποστήριξη κυρίως ε, προς τις ε, οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα ή στην ε, βοήθεια των προσφύγων. Αυτά δεν, θε, δεν θέλαμε να τα περικόψουμε. θέλουμε να μειώσουμε τη γραμμή που αποδημετωπίζεται καταχρηστικά ενδεχομένως από την Τουρκία και δεν ε, λειτουργεί με βάση τις αρχές μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μετά το τομέας 5, ε, εδώ έχουμε 55 εκατομμύρια 27,2 για την Κομισιόν, όχι, 27,8 για την Κομισιόν, 27,2 για τα άλλα όργανα. Για τις ε, συντάξεις και τα ευρωπαϊκά σχολεία δεν πήραξαν τίποτα, αλλά και εδώ θέλω να ρωτήσω πολύ συγκεκριμένα. Τέλος, οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες, εδώ τα, οι πιστώσεις ε, για ορισμένες έχουν περικοπεί στο ΕΚΑ, για παράδειγμα, για την ασφάλεια και την υγεία, το ΣΕΝΤΕΦΟΠ για την επαγγελματική κατάρτιση, για τους σιδηροδρόμους, η Frontex και το Ευρωπαϊκό Γραφείο ε, Υποστήριξης ε, σε Αυτό το ΕΑΖΟ. Ε, εδώ παρουσιάστηκαν δυσκολίες τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχει εξέταση, αλλά αν μπορούμε να τα βάλουμε όλα στο αποθεματικό, είναι αμφίβολο δεν πρέπει να εμποδιστεί πλήρως η εργασία στον ΕΑΖΟ, γιατί αν στο παρελθόν έγιναν σφάλματα, θα πρέπει να φροντίσουμε ούτω ώστε όλα να λειτουργούν ρολόι το 2020. Αλλά ε, δεν θα πρέπει να μειώσουμε τα κονδύλια και να περιορίσουμε το έργο του ΕΑΣΟ το 2020. Αυτό να το διαπιστώσουμε πώς έχει τώρα. Για τα ε, φάρμακα, για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ε, αυτά επίσης θα πρέπει να το δούμε. Μία παρατήρηση επίσης για ιδιαίτερους τομείς, ε, στο, α, το ΣΕΦΙ για την, το Connecting Europe Facility και εδώ 197 εκατομμύρια μείωση. Αυτό αφορά εμβληματικά προγράμματα ε, για την Εσθονία, την Ιταλία, την Ισπανία. Προγράμματα μεγάλα, πολύ σημαντικά και τα οποία τώρα είναι υποσχεδιασμό. Γι' αυτό δεν καταλαβαίνω αυτές τις περικοπές. Θα συζητήσω με το Συμβούλιο και με την Κομισιόν για να δούμε τι επιπτώσεις θα είχε μια τέτοια περικοπή. Για μας, ως ε, γενικός προσανατολισμός, ως γενικό προσανατολισμός, το έγγραφο εργασίας ως εισηγήτρια ε, λέω ότι πρέπει να ακυρώσουμε κάποιες περικοπές που προτείνει το Συμβούλιο και να στηρίξουμε τη θέση της Κομισιόν. Κυρίως όμως ε, αυτό που πρέπει να ε, δούμε στο έγγραφο είναι οι προτεραιότητες για την αλλαγή του κλίματος και για την έρευνα και την καινοτομία. Θα πρέπει επιμείνουμε και στα θέματα της ανεργίας των νέων, εκεί να πούμε τις προτεραιότητές μας, ε, στα πλε... όπως είπαμε για το Εράσμους και αλλού, και τα σημαντικά για την αναπτυξιακή βοήθεια, τα σημαντικά σημεία για τη γνώμη μας. Αυτά είναι οι δικές μας προτεραιότητες, τις έχουμε ορίσει, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, ε, είμαι στη διάθεσή σας για ό,τι ερωτήσεις υπάρχουν. Ε, προσπάθησα να σας κάνω μια επισκόπηση. Θα σας ενημερώνω τακτικά σχετικά με συνομιλίες που θα κάνω και σχετικά με τις ε, συναντήσεις που θα, μια συνάντηση που πρέπει να κάνουμε με τους σκιώδες για να συζητήσουμε πώς θα προχωρήσουμε στρατηγικά ε, απέναντι στο Συμβούλιο. Εγώ δεν θέλω να ε, το επικρίνω το Συμβούλιο, θέλω να είμαι επικοδομητική, αλλά μερικά πράγματα δύσκολα τα καταπίνει κανείς. Και αν ε, μάλιστα δεν παίρνουμε και ερωτη... απαντήσεις στις ερωτήσεις ή να μας λένε κάτι γενικόλογα, ότι θέλουμε να είμαστε προσεκτικοί, να υπάρχει σύνεση. Ε, δεν ξέρω γιατί πρέπει τα περιθώρια να διευρυνθούν. Δεν ξέρω σε τελευταία ανάλυση γιατί το ε, μέσον ευελιξίας δεν αξιοποιείται. Εμείς δεν είμαστε στον πρώτο χρόνο του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου και να μην ξέρουμε. Είμαστε στο τελευταίο χρόνο αυτού του δημοσιονομικού πλαισίου, του πολιετούς. Και δεν καταλαβαίνω. Δεν έχουμε δηλαδή αβεβαιότητες πολλές. Γιατί λοιπόν να κάνουμε τέτοιες περικοπές που θα οδηγήσουν σε, υπο, σε περιορισμό των στόχων μας. Δεν θα φτάσουμε στο στόχο του 20% για το, την αλλαγή του, στα πλαίσια της αλλαγής του κλίματος. Δεν υπάρχει λόγος να μην ε, μένει πιστός στις ειδικέ του τις αποφάσεις του Συμβούλιο. Εμείς υπογράψαμε στο Παρίσι τη Σύμβαση για το κλίμα. Δεν πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε ή στο τομέα της αναπτυξιακής βοήθειας δεν πρέπει να βάλουμε προτεραιότητες για να βοηθήσουμε τις χώρες που χρειάζονται. Δηλαδή δρά πολύ τεχνοκρατικά το Συμβούλιο και λυπάμαι πολύ γι' αυτό. Εγώ θέλω να είμαι επικοδομητική. Αν μπορούμε και έχει νόημα να κάνουμε κάποια περικοπή και αν τα χρήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν καλύτερα αλλού, ευχαρίστω. Αλλά στα τυφλά περικοπές έτσι καθαρά τεχνοκρατικά, τα οποία βλάπτουν την ουσία των θεμάτων, αυτό εγώ δεν το δέχομαι ως εισηγήτρια. Ξανά σας ευχαριστώ όλους θερμά. Ευχαριστώ κυρία Χολμάιερ. Ισκιώδης τώρα. Ο κύριος Λάρου Τουρού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την εισηγήτρια εκ μέρου των Σοσιαλδημοκρατών. Πρέπει να πω ότι συμμεριζόμαστε πολλέ από τι ανησυχίε ε, και από τι ερωτήσει σα. Πρέπει να καινοτομήσουμε, να επενδύσουμε και όχι να μειώσουμε τον προπολογισμό. Είμαι νέος βουλευτής ε, και όπως πολλοί από εσάς έτσι και εγώ χάρηκα με τη μεγάλη προσέλευση σε ευρωεκλογέ. Ε, περισσότεροι είχαμε υποσχεθεί αλλαγή της Ευρώπης. Ε, δεν το επιτρέπει όμως αυτό ο προϋπολογισμός όπως προτείνεται. Είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. Είδαμε τεράστια προβλήματα φέτος και οι ασφαλιστικές εταιρείε μας δείχνουν πώς αναπτύσσεται το κόστος ε, βλέπουμε δηλαδή ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν δημοσιονομικές επιπτώσεις ε, και μάλιστα 2,5% ε, επί 2,5% έχουν πολλαπλασιαστεί και στις νότιες χώρες ε, είναι πολύ περιορισμένοι οι ασφαλίσεις ε, και τεράστιες καταστροφές. Κύριε Φοντερ είπε ότι η προτεραιότητα της είναι η κλιματική αλλαγή. Το επικροτήσαμε αυτό και είπε για τις 100 πρώτες ημέρες. Αλλά πώς θα έχουμε επιτάχυνση σε αυτό το μέτωπο εάν μειώνονται τα μέσα τα χρηματοδοτικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι αν θέλουμε να είμαστε στο ύψο των ε, απαιτήσεων ε, θα έπρεπε να έχουμε περισσοτερε περισσότερε Αλλά λείπουν 170 με 290 δι ετησίω Αυτή είναι η τελευταία έκθεση του Νοεμβρίου και στον προτινόμενο προπολογισμό, η αύξηση του προπολογισμού για το επόμενο έτος είναι μόνο 0,4 δι. Μόνο 0,4 δι. Αν ληφθεί υπόψη και ο πληθωρισμός δεν είμαστε στο ύψο ε, των προκλήσεων που έχουμε να αντιμετωπίσουμε μέσα στι 100 πρώτε μέρε, λέει η κυρία Φοντρελάιν, πώ θα βοηθήσει τα κράτη-μέλη για τι συγκοινωνίε, τι δημόσιε, την ενεργειακή απόδοση. Δεύτερον, Μάλλον σίγουρα το 2020 θα έχουμε μία νέα χρηματοπιστωτική κρίση. Βλέπουμε το δημόσιο και ιδιωτικό χρέος της ΕΙΠΑ ε, το συνολικό χρέος τους αυξήθηκε κατά 2,530 δις ε, στη ΣΥΠΑ. Ε, είναι κάτι το οποίο ξεπερνάει και το ΑΕΠ της Γαλλίας. Και λέει και το Δέλτα Νιτάφ ότι θα έχουμε νέα δημοσιονομική κρίση. Το βλέπουμε ε, και σε κάποιες εφημερίδες, βλέπουμε κερδοσκοπία τρομερή. Το 2017 είχε φτάσει στα 14.000, ε, μετά ανέβηκε ακόμη περισσότερο, έχει φτάσει και στα 26.000, 26.000 πόντους ε, το το Dow Jones. Κρίση μεγάλη θα έχουμε και είπε και η Κριστίν Λαγκάρντι, η Ευρώπη δεν είναι έτοιμη για μια νέα τέτοια κρίση. Πώς θα επηρεάσουν όλα αυτά λοιπόν τον προπολογισμό μας. Είμαστε πάρα πολύ ευάλωτοι. Και έχουμε τις προβλέψεις του ΔΕΛΤΑΝΤΑΦ και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Ε, εμείς θέλουμε να εφαρμόσουμε την ευελιξία και να αξιοποιήσουμε για τους νέους, για το έρασμος, ε, ως το δυνατόν αυτό το μέσο. Θέλουμε να ε, μην γίνουν πράξει περικοπές που προτείνει το Συμβούλιο, αλλά πρέπει να αξιοποιήσουμε και νέα εργαλεία, ε, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να έχουμε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της κλιματικής και κοινωνικής κρίσης το επόμενο ΠΔΠ. Ποια είναι αυτά τα εργαλεία ε, σε ό,τι αφορά την ασπίδα για την απασχόληση. Κύριε Φοντερλάιν θέλει να υπάρχει ένα σύστημα αντασφάλισης για την ανεργία και σίγουρα πρέπει να βοηθηθούν τα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση του φαινομένου της ανεργίας. Μίλησε όμως ε, ε, και για ένα γερμανικό σύστημα η κυρία Φοντριλάιεν. Είναι ένα σύστημα που εφαρμόστηκε το 2009 στη Γερμανία. Μειώθηκε ο χρόνος εργασίας και όχι το προσωπικό και το 98% ε, το κράταγε. Αυτό το σύστημα ε, ωφέλησε πάνω από ένα εκατομμύριο του στη Γερμανία που διατήρησαν τη δουλειά τους. Και ο πρόεδρος Κέννεντι, αν θυμάστε, έλεγε ότι αν υπάρχει ε, ήλιος ε, θέλουμε να επισκευάσουμε τη στέγη για να προστατεύσουμε. Πρέπει λοιπόν εμείς αυτό να κάνουμε, να επισκευάσουμε τη στέγη του κοινού αυτού οίκου ε, για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ανεργία. Και ο Ζακ Ντελόρ πριν από 20 χρόνια έλεγε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί το κοινωνικό και φορολογικό ντάμπινγκ. 45% ήταν ο φόρος των κερδών των επιχειρήσεων, 19% είναι τώρα. Και θέλουμε όλη η φορολογική δικαιοσύνη. Πρέπει λοιπόν να λυθούν αυτά τα προβλήματα ε, και είναι μια προϋπόθεση. Εμείς θα το θέσουμε ως όρο στην ομάδα μας ε, για τα επόμενα έτη να έχουμε δηλαδή νέες μεθόδους χρηματοδότηση για τον ε, επόμενο πολιετές μασιομικό πρόγραμμα. Δεν μπορούσα να μακρηγορήσω ακόμη περισσότερο, αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ως ομάδα για αυτό το θέμα στο επόμενο ΠΔΕΛΤΑΠΗ. Bonjour. Καλημέρα. Προέρχομαι από την ε, Ρουμανία και ευχαριστώ την εισηγήτρια και το επιτελείο της για αυτήν την ε, πάρα πολύ ενδελεχή εργασία τα συζητήσαμε και θα σας πούμε την αρχική μας τοποθέτηση. Έχουμε την ίδια προσέγγιση όπως έχει και η κυρία Μονίκα Χόλμαγερ. Έχουμε βεβαίω συγκεκριμένες προτεραιότητες, ορίζον 2020 που υπέστη την μεγάλη περικοπή για το κλίμα, 20% ε, αλλά θέλουμε να υπάρξει καινοτομία στην οικονομία για να προστατευτεί το περιβάλλον. Επίσης, είπαμε ότι ολοκληρώνεται τώρα το πολιτές πλαίσιο, οπότε θα πρέπει να γίνει απορρόφηση από τις χώρες και να σταματήσει ε, αυτό το χάσμα Ανατολής Δύσης. Οπότε να ολοκληρωθεί η διαδρομή αυτού του πολιτής πλαισίου με επιτυχία τεχνική αρρωγή και έχουμε μια άριστη έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολισμού του Μαρτίου του 19 κύριε Χολμάγερ και λέει ότι η τεχνική αρρωγή είναι πάρα πολύ σημαντική ούτως ώστε να έχουμε ε, σωστή πολιτική συνοχή. Οπότε εμεί θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε και επίσης και, ε, γίνει κάτι και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κύριε Αντρίσεν. Ευχαριστώ κυρία Χόλμαγερ για την έκθεσή σας. Συμφωνούμε σχεδόν 100%. Επίσης οι πράσινοι έχουμε σοκαριστεί από την τοποθέτηση του Συμβουλίου. Αν κανείς ακούσει ακριβώς τι λέει η Φιλανδική Προεδρία και κατόπιν μελετήσει τα έγγραφα, θα, θα δει ότι είναι μέρα με τη νύχτα. Πολλά προβλήματα να μην επαναλάβω όλα αυτά που ήδη αναφέρθηκαν, αλλά για μας το βασικό θέμα είναι η κλιματική αλλαγή και όχι μόνο δεν τηρούμε το σύστημα στο Παρίσι, αλλά δεν έχουμε φτάσει ούτε το 20% σε σχέση με τον προϋπολογισμό. Οπότε θα πρέπει όχι μόνο τον προπολογισμό να επιστατεύσουμε για τη συμφωνία ε, των Παρισιών, αλλά και να κάνουμε κάτι για να πετύχουμε το 20%. Αυτό έχει, έχει προκύψει φάσεις διαφόρων οργάνων, εκτό από το Συμβούλιο. Άρα θα πρέπει να έχουμε κάποια στροφή στη στάση μας στις διαπραγματεύσεις επόμενες εβδομάδες. Κάτι άλλο τώρα, κανείς δεν το ανέφερε. Αλλά είναι σημαντικό για την νεολαία και την απασχόληση και το σχετικό ε, μέσο ε, πολιτικής απασχόληση ε, για τους νέους. Χρειάζεται να βοηθήσει περισσότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί υπάρχουν περικοπές στα σχετικά προγράμματα. Για να το ξαναδούμε. Το είπαν και οι σοσιαλιστές εν ώψη της οικονομικής συγκυρίας τα μέσα επόμενα χρόνια. Τα πράγματα θα χειροτερέψουν αν δεν κάνουμε τίποτα. Ε, γι' αυτό και εμείς θεωρούμε ότι πρόκειται για κάτι πολύ σημαντικό. Πρέπει να το λάβουμε υπόψη για την χρήση του 20 στον προπολογισμό. Θα τα δούμε τι αμέσως εβδομάδες γιατί πρέπει να γίνουν σημαντικές αλλαγές. Να υπενθυμίσουμε στο Συμβούλιο το τι λέει, τι υπόσχεται στα κρατημέλη. Γερμανία, Σκανδιναβία. Όλοι όλοι υπόσχονται δαπάνες υπέρ του κλίματος, αλλά πούντες. Κυρία Λαπόρτ, Συνάδελφοι, θεωρούμε ότι είναι σωστή η θέση του Συμβουλίου για τον προϋπολογισμό του 20. Θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με την Εθνική Οικονομική Πολιτική και το Συμβούλιο. Έχουμε την πρόταση επομένως, αλλά θα πρέπει να τροποποιηθεί πρώτα-πρώτα για την προένταξη θεωρούμε ότι θα πρέπει να σταματήσει η επάπειρον διεύρυνση της Ένωσης. Υπάρχουν και σημαντικά προβλήματα. Θα δούμε τι θα γίνει με τον τουρκικό εκβιασμό για το μεταναστευτικό. Αλλά θα, αφού έχουμε ένα όργανο προστασίας των συνόρων, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους ε, Τούρκους και όχι στην Frontex. Επίσης για τις διαρθωτικές ε, μεταρρυθμίσεις εμείς είμαστε κατά τα κράτη-μέλη ε, δυσκολεύονται να εφαρμόσουν τις συστάσεις της Κομισιόν. Εμείς έχουμε πρόβλημα όσον αφορά τα επιδόματα ανεργίας και ε, απειλεί η Επιτροπή να μας κλείσει τη στρόφιγγα εάν δεν κάνουμε αυτά τα οποία έχουμε δεσμευθεί. Πρόκειται για εκβιασμό. Επίσης, οι ανακοινώσεις της Ένωσης είναι σαν προπαγάνδα. Δεν βελτιώνει την καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων. Ουσιαστικά τα έργα χρηματοδοτούνται από τα κράτη-μέλη, από τι εθνικέ οικονομίε και συγκεκριμένα από του ε, φορολογουμένου, του Γάλλου φορολογουμένου. Ε, ε, Ευχαριστώ. Εγώ Μιλώ εκ μέρους των συντηρητικών. Σύντομα λοιπόν, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι υπήρξαν πολλά κράτη τα οποία άσκησαν κριτική στο Συμβούλιο και αν δει κανείς τις προκλήσεις ε, που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τις δράσεις που θέλουμε να φέρουμε σε πέρα, σίγουρα όλα αυτά είναι ανησυχητικά. Εγώ είμαι νέο ευρωβουλευτή, έχω δει όμως πολλά πράγματα στο δικό μου κοινοβούλιο, το εθνικό, και πρέπει κανείς να διερωτηθεί ποιος εκπώνησε τη θέση αυτή ε, στο πόδι, έγινε ε, κάποια αυτοσχεδίασαν, ε, δεν φαίνεται να είναι κάτι που είναι αποτέλεσμα όρημη σκέψης αυτό το σχέδιο προπολογισμού. Uh, Κύριο Χάουρ, ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν κάποιοι οποίοι λένε ότι είναι καλό να ανεβαίνει ο προϋπολογισμός. Ε, αυτό είναι ανοησία και αυτό αποδεικνύεται αν δει και τα στοιχεία ε, του προεπολογισμού για φέτος, που ουσιαστικά είναι μια αυτή γραμμή και ε, υπάρχουν κάποιες περικοπές, βέβαια, που προτείνονται από το Συμβούλιο είπε πολύ εύγλωτα ο προλαλής σας συνάδελφος όμως ότι είναι ρηψοκίνδυνη και αρνητική δυνητικά η προσέγγιση αυτή. Βέβαια, το πρόβλημα δεν είναι ε, ο προπολογισμό και τα ποσά, τα ονομαστικά, αλλά ότι δεν υπάρχει ε, συνέχεια και λογική δεν υπάρχει λογική προσέγγιση σε σχέση με το σχέδιο αυτό του προπολογισμού της, ε, του Συμβουλίου. Γιατί δεν έχει και καμία σχεδόν σχέση με τις προτεραιότητες που είχε ήδη θέσει για την Ευρωπαϊκή Ένωση το Συμβούλιο. Έχουμε στο 1α περικοπές ε, που πραγματικά έρχονται σε αντίθεση με τα όσα έχει πει το Συμβούλιο. Δεν έχει νόημα, για παράδειγμα, οι ε, επενδύσεις ε, στην έρευνα για το κλίμα που ε, εγκρίναμε με το δεύτερο διορθωτικό επεπολογισμό να αυξάνεται αυτές οι δαπάνες και να μειώνει το επόμενο έτος. Θα κάνουμε τροπολογίες. Ε, αλλά τα πράγματα φαίνεται να πηγαίνουν χειρότερα. Επίσης, είμαι και ηγητής σε μια επιτροπή και έκανε τη σχετική γνωμοδότηση, σίγουρα η η αγορά είναι μια προτεραιότητα και το λένε επανειλημμένο στα κρατημέλη και όποιοι έρχονται εδώ. Και πάλι όμως έχουμε πρόταση περικοπών. Και αυτό δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την πρόοδο που λένε ότι θέλουν και ότι είναι προτεραιότητα οι χώρες μέλη του Συμβουλίου. και δεν υπάρχει χρηματοδότηση για την ε, απασχόληση για την νεολαία, δεν θα ε, πάψει να εμφίσταται αυτό το πρόβλημα. Το πρόγραμμα είχε επενδύσεις και επιτυχίες, αλλά ε, δεν είναι ένα πρόγραμμα αυτό που μόνο για την κρίση δημιουργήθηκε και θα πάψει να υφίσταται, αλλά είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα συνεχίσει να υφίσταται λόγω και αλλαγών στη φύση της αγοράς εργασίας, της διάθεσης αγοράς εργασίας και των, α, απασχόλησης. Και σίγουρα θα επηρεάζει τους νέους όλο και περισσότερο ε, η διάρθρωση της ε, αγοράς απασχόλησης μέχρι ότι υπάρξει μια αναδιάρθρωση και είναι πιο φιλική προς τον εργαζόμενο. και είναι κοντόθωρη, άκρος κοντόθωρη προσέγγιση του Συμβουλίου σε αυτούς τους τομείς. Αν όμως δει κανεί τι τεχνικές λεπτομέρειες των εγγράφων, εκεί αντιλαμβάνεται πλήρως ε, την ασυνέπεια και την αντίφαση. Να δούμε τι γίνεται για να πάρω μια αναλογία για τη χορτικοπτική ε, μηχανή τι γίνεται στον τομέα IT, πληροφορικής. Δεν ξέρω. Έχουν διαρρέσει με κατά 25-26 και έχουν ξηρίσει, έχουν ε, ε, κάνει αυτές τις γραμμικές ε, περικοπές. Δηλαδή αναζητούν ένα μηχανισμό απλά για ε, γενικές περικοπές τύπου χορτοκοπτικής μηχανής, χωρίς καμία μελέτη του αν κάτι αποδίδει δεν αποδίδει. Και όλα αυτά νομίζω δείχνουν πόσο ανεπαρκή είναι η διαδικασία και η προσέγγιση αυτή. Τέλος, για τη Frontex και τις προτινόμενες εκεί περικοπές εγώ άσκησα δερμία κριτική για τον τρόπο με τον οποίο ε, έχουμε αντιδράσει μετά την ανακοίνωση του Γιούνκερ για τις προθέσεις του για το επόμενο ΠΔΠ. Δεν βλέπω να έχουμε ούτε εδώ συνέπεια, ε, συνεκτική στάση σε σχέση με τις προτάσεις για το επόμενο έτος. Θέλουμε λοιπόν όχι απλά να αναστρέψουμε αυτές τις περικοπές, αλλά να δώσουμε και μία λογική σε αυτό τον προπολογισμό. Ευχαριστώ κύριε Σμουρεσάν, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να προσθέσω κι εγώ κάτι. Αυτό που βλέπουμε είναι το business as usual. Τα ίδια κάνει κάθε χρόνο. Μιλάμε για προτεραιότητες πρώτα και ως κοινοβούλιο εμείς ε, προσπαθήσαμε να βρούμε τη σωστή χρηματοδότηση για τις προτεραιότητες. Ε, το Συμβούλιο λέει η ασφάλεια, το κλίμα ε, είναι, ε, και πολλά άλλα είναι σημαντικά, αλλά κάνει περικοπές ταυτόχρονα. σημαντικό είναι να είμαστε ενωμένοι. Η θέση της εισηγήτριας της διαπραγματεύσεις, στις συνομιλίες με την Κομισιόν μας έχει πίσω τις ενωμένους. αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, το 2020 είναι η τελευταία χρονιά του τωρινού πολιετούς. Στην αρχή των πολιετών πιέζονται τα ε, κράτη-μέλη να διαθέσουν χρήματα. Θα πρέπει και τώρα να πιέσουμε τα κράτη-μέλη για ένα σωστό προϋπολογισμό που θα ωφελεί τα κράτη-μέλη. Και στο τέλος θα στο τέλος του πολιετούς θα πρέπει να πιέζομαι τα κράτη-μέλη να καταβάλουν στον προϋπολογισμό ε, ανάλογα με τις υποχρεώσεις τους. Δύο, δύο φορές τους πιέζουμε. Ε, στην αρχή και στο τέλος. Τώρα είμαστε στο τέλος του, αυτού του πολιετούς και διαβάζοντας τη θέση του Συμβουλίου βλέπουμε ότι τώρα η προτεραιότητα είναι να διασφαλίσει ε, περιθώρια. Απαράδεκτο, γιατί η προτεραιότητα του προϋπολογισμού κατά τη γνώμη μου είναι να εντοπίζει τι περιμένει ο κόσμος από την Ευρώπη, να διαθέτει τα, κατάλληλα κονδύλια και να διασφαλίσει ότι δαπανώνται σωστά. Δεν μπορεί να είναι προτεραιότητα να μην δαπανάτε ο προϋπολογισμός, δεν είναι προτεραιότητα αυτή και να έχουμε περιθώρια. Ένα υψηλό περιθώριο δεν έχει νόημα ε, στο τελευταίο χρόνο του πολιετούς. Ε, πάντα λοιπόν λέω στην αρχή το περιθώριο θα πρέπει να είναι υψηλό γιατί υπάρχουν απρόβλεπτα. Ποιος ξέρει τι μπορεί να γίνουν μέσα σε 7 χρόνια. Ε, είχαμε γιατί πολλά απρόβλεπτα το Juncker 1, Juncker 2, Αφγανιστάν, το, ε, Τουρκία και όλα τα απρόβλεπτα Στο τέλος όμως δεν μπορεί, τι μπορεί να συμβεί γι' αυτό πρέπει να είναι μικρότερο το περιθώριο. Το επιχείρημα για μεγάλα περιθώρια είναι ασθενέστερο από ποτέ. Τέλος, η συμμετοχή στις ευρωεκλογέ ήταν υψηλή, ο κόσμος ήρθε να ψηφίσει, ήθελε να βοηθήσει η Ευρώπη για την ασφάλεια, την αλλαγή του κλίματος, ε, τη γενοτομία ε, και τι βλέπει το Συμβούλιο. Για τους νέους ε, κόβει το μέσον για την, αυτή την πρωτοβουλία για την ενεργεία των νέων ή κόβουν το εσωτερικής ασφάλειας στο ταμείο και, άλλα τα ταμεία. Ε, αυτοί που θέλουν να αντιμετωπίσουν την νόμιμη μετανάστευση και εκεί κόβουν το αμύφ κατά 35 εκατομμύρια ευρώ. Όλο περίκοπες για τη φτώχεια στις τρίτες χώρες. Εδώ 70 εκατομμύρια. Ε, για να, γιατί θεωρούν φαίνεται ότι είναι καλά τα πράγματα στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Τι θέλω να πω. Αυτές οι περικοπές είναι γελίες. Γι' αυτό το 2018 που ήμουν γενικό συζητητή για τον προϋπολογισμό της Ένωσης δεν ασχολήθηκα να μιλήσω για αυτές τις περικοπές στη διαπραγματεύση. Είπα τις απορρίπτουμε. Είχαμε μεγάλη πλειοψηφία υπέρ της απόρριψης των περικοπών και είπα μετά θα συζητήσουμε να δούμε πού χρειάζονται περισσότερα κονδύλια. Γι' αυτό πιστεύω και το λέω στην εισηγήτρια ότι τη συμβουλεύω να μην μιλήσει πολύ για τις περικοπές, να συμφωνήσουμε ότι είναι γελίες, τις απορρίπτουμε, πάει και τέλειωσε και μετά θα πρέπει να αρχίσει μια έλογη συζήτηση για το τι πρέπει να γίνει. Τέλος, αυτός είναι ο πρώτος χρόνος της θητείας μας στο Κοινοβούλιο. Ε, το παρακολουθούν όλοι πολύ. Αν φερθούμε αδύναμα τώρα, αυτό θα μας σημαδέψει για την υπόλοιπη θητεία και ο... στο... δεν έχετε αποφασίσει οι σοσιαλιστές για τον... Ποιος είναι ο συνεισηγητής του Γιάν Ε, ο Γιάνν είναι σίγουρος μέχρι στιγμής. Εντάξει. Αν υποχωρήσουμε τώρα θα μας θεωρούν αδύναμους για το υπόλοιπο της θητείας και θα είναι και η διαπραγματευτική μας θέση αδύναμη για το πολιετές δημοσιονομικό. Να είμαστε ενωμένοι και να είμαστε ισχυροί στην αντιπαράθεση με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Σαφές. Ο κύριος Φερνάντες. Ευχαριστώ πρόεδρε. Συγχαρητήρια στην ε, εισηγήτρια και χαίρομαι για αυτό το πνεύμα, την ατμόσφαιρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση που το χρειαζόμαστε για να έχουμε ένα αξιόλογο προπολογισμό του 2020. Πολύ σημαντικό γιατί θα αποκτήσουμε το 20 και το νέο δημοσιονομικό πολιτες πλαίσιο να δούμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς από το 2020 κιόλας θα μπορέσει να τάξει τις νέες της προτεραιότητες τα λοιπά, business as usual. Και αν κάποια μέρα το κοινοβούλιο πει στο Συμβούλιο, καλώς, ό,τι πείτε για τον προϋπολογισμό, το Συμβούλιο θα μας απαντήσει, για περιμένετε, γιατί υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να τα αλλάξουμε και να τα βελτιώσουμε. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Γιατί πάντα τα ίδια. Ρολέτα. Υπάρχουν κάποια κονδύλια, κάποια, κάποια τα κόβουν για να πάνε στο 1% των πιστώσεων πληρωμών. Ε, αυτό είναι το πνεύμα του, η λογική τους. Κόβουν όπου να είναι και περιμένουν εμείς να λάβουμε τι ευθύνες μας. Θεωρούν ότι εμείς έχουμε την ευθύνη για να κάνουμε κάποια πρόταση, ενώ εκείνοι κόβουν ό,τι να είναι. Αυτά για να μην χάνουμε χρόνο σε σχέση με το που έχουν κόψει και έτσι κι αλλιώ ε, βρίσκονται σε κάποια αντίφαση, γελία. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Αλλά εμείς θα είμαστε σοβαροί ως συνήθως. Και σας τονίζω το εξής. Έχουμε την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων που εκεί δεν είναι απλώς μια ρουλέτα για τα κράτη-μέλη. Γίνεται ε, τυχαία ε, εδώ η περικοπή γιατί έτσι, γιατί έτσι έτυχε. Αλλά στα πλαίσια της πρωτοβουλίας τα κράτη-μέλη καλύπτουν τον προπολογισμό το μισό και το άλλο μισό προέρχεται από την εταιρική συμφωνία των διαθετικών ε, ταμείων και τα κράτη-μέλη δεν θέλουν να αλλάξουν αυτή την συμφωνία εταιρικής σχέσης και λένε θα γίνει γραφειοκρατικά, θα έχουμε καθυστερήσει. Θα πρέπει να ζητηθεί από τα κράτη-μέλη να μειώσουν τη σχετική γραφειοκρατία, διότι δεν είναι δυνατόν να δεχθούμε κάτι τέτοιο για την ε, πρωτοβουλία. Γιατί έτσι θα φυγούν και οι εταιρικές συμφωνίες κάθε κράτους μέλους. Αυτό ήδη το έχουμε δει, έχει συμβεί στο παρελθόν. Με την πρωτοβουλία τα μισά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα άλλα μισά από τα διορθωτικά ταμεία, από το κοινωνικό ταμείο δηλαδή. Και θα πρέπει εμείς να τους εξωθήσουμε σε μεταβολές, οι οποίες όμως να είναι γρήγορα ε, διεκπεριωμένες. Και, με κατακλείδη, ο προϋπολογισμός αφορά όλα τα κρατημέλη. Όλοι ωφελούνται. Ακόμα και εκείνοι που εισφέρουν περισσότερα και με το 1% του εθνικού ΑΕΠ ε, έχουμε μία πάρα πολύ μεγάλη προσθέμενη αξία. Και βέβαια με το 1% δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν όλες οι προκλήσεις. Να γιατί πρέπει να ενισχυθεί. Αυτός ο προηγούμενος που δίνει τόσο μεγάλη προσθέμενη αξία. Ο πρόεδρος. Είναι το λόγο στον επόμενο. Κυρίες και κύριοι, η εισηγήτρια Χολμάιερ και η Σκιώδης είπαν πολύ ωραία πράγματα. Φαίνεται ότι το Συμβούλιο θέλει να μας στείλει το μήνυμα ότι τέλειωσαν οι κρίσεις σας, άσυλο, μετανάστευση, απασχόληση των νέων, κλιματική αλλαγή κυρίως, ότι λήξανε, λήξανε τα θέματα αλλά το μήνυμα πριν από το καλοκαίρι ήταν διαφορετικό. Η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν μίλησε πολύ για το κλίμα και εμεί ε, όταν την εγκρίναμε μίλησε για το κλίμα που θα μετριάσει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, για προγράμματα επενδύσεων, όλα αυτά σημαίνουν χρήμα, σημαίνουν 20% του προϋπολογισμού τα επόμενα έτη, αν όχι και παραπάνω τώρα μετά το καλοκαίρι έρχονται και δίνουν άλλο μήνυμα ότι όλα αυτά τα μέσα μειώνονται. Αυτό είναι πάρα πολύ ε, διαφορετικό μήνυμα. Είναι σε παραφωνία με τα προηγούμενα. Τώρα, για το 2020, η μείωση της πρωτοβουλίας για την ε, απασχόληση των νέων είναι παράλογη. Ε, πολλοί στην προεκλογική, στις προεκλογικές του εκστρατείας μίλησαν για αυτά τα θέματα ε, ε, με τους νέους, μίλησαν ε, με αυτούς και είδαν ότι... Και, ε, ότι η κρίση δεν έχει τελειώσει, άρα τα χρήματα χρειάζονται. Τώρα, ο προϋπολογισμός συζητήθηκε πριν από το καλοκαίρι το Συμβούλιο, γιατί αν παρακολουθήσαμε το, το τι γινόταν το καλοκαίρι, εκεί ήταν μια περίοδος κρίσης. Έχουμε όλες τις κρίσεις και από την άλλη βλέπουμε όμως τώρα ότι έχουμε περικοπές. Τέλος, δεν είναι μόνο το Συμβούλιο που κάνει τις περικοπές, θα πρέπει να δούμε και τι κάνει η Κομισιόν. Πιστεύω... Ε, για στα πλαίσια του Ρινιού το γεγονός ότι μειώθηκε και ο μηχανισμός πρόληψης ε, είναι τρέλα. Η Αμαζονία μπορεί να περιμένει, φαίνεται ε, να είναι το μήνυμα που στείλανε. Θα πρέπει λοιπόν να αναμένουμε ε, διόρθωση αυτής της θέσης. Παλιά στη χώρα μου, την Πολωνία, έλεγαν ότι μπορούμε να προβλέψουμε μια πυρκαγιά στο σπίτι μας και μετά να βάλουμε εμείς η ίδια τη φωτιά. Ε, αυτό σήμαινε καλή πρόβλεψη. Σαν να λέμε ότι προβλέπουμε ότι αυτό το σπίτι θα πάρει φωτιά και μετά βάζουμε φωτιά στο σπίτι αυτό. Η θέση του Κοινοβουλίου στη συζήτηση για τα πολιετή δημοσιονομικά πλαίσια και συμφωνώ με τους Μωρισάν και Φερνάντες, εμείς λέμε στη θέση μας ότι χρειαζόμαστε περισσότερα κονδύλια στον προϋπολογισμό ή χρειάζεται να μεγαλώσει ο προϋπολογισμός λόγω των σημαντικών νέων προκλήσεων. Υπάρχουν κάποιοι, κάποιες κυβερνήσεις και κάποιες συνάδελφοι που λένε όχι. Όχι λένε, δεν χρειάζονται όλα αυτά τα παραπάνω. Και τώρα προχωρούν σε περικοπές. Τι σημαίνει αυτό για τις επόμενες συζητήσεις για το πολιετές. Ε, θέλουν να αποδείξουν ότι δεν χρειάζεται. Ότι ο προπολογισμό είναι πολύ μεγάλος. Βέβαια μπορούμε να πούμε όχι. Να πούμε όχι είναι παρά, παράτυπα όλα αυτά, ε, παράλογα κλπ. Αλλά πρέπει να προχωρήσουμε παραπέρα και να δούμε γιατί προτείνεται τις περικοπές. Ξέρουμε ότι δεν είναι λογικό αυτό, αλλά πρέπει να κάνουμε την ερώτηση επειδή δεν, μπορούμε, μπορούν να δαπανηθούν τα κονδύλια ή επειδή τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να τα δαπανίσουν τα κονδύλια ή επειδή το πρόγραμμα ήταν πολύ μεγάλο. Γιατί αν είναι πολύ μεγάλο χρειαζόμαστε λιγότερα στο νέο πολιετές. Θα πρέπει να προχωρήσουμε λογικά, να δούμε ε, τα, ε, ότι ε, χρειάζονται χρήματα. Η ερώτηση, λοιπόν, το πραγματικό ερώτημα είναι γιατί δεν, δαπανάτε το, το, δεν δαπανώνται τα κονδύλια. Γιατί δεν τα καταφέρνει η Κομισιόν, δεν τα καταφέρνουν οι κυβερνήσεις ή δεν ε, υλοποιείται καλά το πρόγραμμα. Πρέπει να απορρίψουμε τη θέση, αλλά δεν πρέπει να σταματήσουμε εκεί. Θα πρέπει να, δούμε, να, ρωτήσουμε τι έγινε. Αλλιώς ε, αποδυναμώνεται το επιχείρημά μας και θα έρθουν και θα μας πούνε «Συγγνώμη, ε, με αυτές τις περικοπές το 1,3 είναι, το, ε, είναι ε, ελάχιστο, το 1,0 είναι καλύτερο. Και εμείς λέμε όχι γιατί πιστεύουμε ότι είναι λάθος. Θα πρέπει όμως να εντοπίσουμε και το λάθος και ποιος είναι υπεύθυνο γι' αυτό, δηλαδή για τη μη σωστή διάθεση των κονδυλίων. Δεν πρέπει να είμαστε απλουστευτικοί και να πούμε όχι, σκέτα, ναι, ναι τα σκέτα, όχι μεν, αλλά δώστε μας σαφείς εξηγήσει σχετικά με το τι γίνεται. Ευχαριστώ. Άλλα σχόλια από το Κοινοβούλιο. Και εγώ να πω κάτι. Μετά την πενταετή μου πήρα ως υπουργό Οικονομικών που συζητούσαμε για προγράμματα. Νομίζω ότι είναι πολύ κακή πολιτική να μην εξηγούμε τι κάνουμε. Αυτό που λέγατε πριν από λίγο. Η κλιματική αλλαγή είναι σημαντική προτεραιότητα. Μπορεί να υπάρχουν παρόλα αυτά κάποια ε, επιχειρήματα υπέρ της περικοπής κάποιων προγραμμάτων για την κλιματική αλλαγή. Οκ, okay, μπορεί να ισχύει αυτό. Αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν υπάρχει αντίφαση αφενός ε, ότι, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για το κλίμα και να κάνουμε κάτι και από την άλλη να εντοπίζουμε δυναμίες στα υφιστάμενα προγράμματα. Αυτό μπορεί να γίνει. Δεν είναι ασύμβατα τα δύο. Αλλά η εξήγηση, η αιτιολόγηση είναι πάντα σημαντική. Δεν μπορεί να περικόπτουμε τον προϋπολογισμό σε αυτό σκοπό. Ε, πρέπει να αιτιολογούμε λοιπόν. Γιατί γίνεται αυτό που γίνεται. Και προφανώς σε ευρωπαϊκό επίπεδο χρειάζεται αυτό ε, για ένα λόγο παραπάνω, γιατί προτείνονται περικοπές. Θέλετε να μιλήσετε. Πολύ γρήγορα. Δεν ήθελα να πάρω το λόγο γιατί συμφωνούσα και σε πολύ μεγάλο βαθμό με όσα επιχειρήματα αναφέρθηκαν αλλά η δική σας παρέμβαση με έκανε να αντιδράσω και εσείς στα πέντε χρόνια στο Συμβούλιο και σίγουρα είναι όλα αυτά που λέτε πολύ σημαντικά. Συμφωνώ ότι μπορεί κάποια προγράμματα να μην λειτουργούν. Να, ναι, μπορεί να συμβεί αυτό. Όμω, δεν αφαιρείται ε, τα κονδύλια από τα προγράμματα. Δεν κάνουμε έτσι. Αυτό που κάνουμε είναι να βελτιώσουμε τα προγράμματα. Παραδείγματο χάρη, κλιματική αλλαγή. Α πούμε ότι έχουμε ένα πρόγραμμα που δεν ε, πληρεί. Ε, τι κάνει το Συμβούλιο, δεν λειτουργεί το πρόγραμμα, παίρνουμε τη χρηματοδότηση και το πετάμε στα σκουπίδια. Εμεί ω Κοινοβούλιο πώ λειτουργούμε, βελτιώνουμε το πρόγραμμα γιατί είναι ανάγκη να παραμείνει και δεν κόβουμε τη χρηματοδότηση πρέπει να ζητήσουμε εξηγήσει από το Συμβουλίο. Είπατε, μα τις έχουμε ακούσει και πραγματικά δεν έχουν λογική. Γιατί αν δείτε τι λένε, επενδύσει, καινοτομία, κλιματική αλλαγή είναι προτεραιότητε. Και μετά τι κάνουν, περικόπτουν προγράμματα που δεν έχουν υψηλό ποσοστό απόρροφηση. Μα δεν είναι σωστό αυτό. Στον ορίζοντα 2020 το 90% των προγραμμάτων τα απορρίπτουν, όχι γιατί είναι καλά, αλλά γιατί ε, δεν έχουν ε, χρήματα. Επίση, ε, έχουμε άλλα προγράμματα τα οποία συμφω... λειτουργούν πολύ καλά. Και ένα από αυτά είναι η, το πρόγραμμα για την ανεργία των νέων, που είναι ένα δομικό πρόβλημα, δεν είναι κάτι περιστασιακό. Άρα και οι λόγοι που προβάλλουν, τα επιχειρήματα τα οποία αναφέρουν, Ακόμα και αν θέλαμε να μπούμε στη θέση του Συμβουλίου και να λάβουμε υπόψη αυτά τα κίνητρα, ούτε πολιτικό ούτε οικονομικό θεμητό κίνητρο υπάρχει. Οι Υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών το μόνο που θέλουν να κάνουν είναι να σώσουν ό,τι μπορούν για να μην δίνουν κονδύλια στην Ευρώπη. Ας το πούνε όμως και να μην λένε δικαιολογίε ότι δεν υπάρχει απορρόφηση, δεν είναι απαραίτητο το πρόγραμμα, δεν λειτουργεί κτλ θέλουν 1% για τις πληρωμές και αυτό είναι το μόνο το οποίο προσπαθούν να επιτύχουν με οποιαδήποτε άσχετα επιχειρήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Χολμαϊερ, να σας δώσω... Όχι, να διευκρινίσω κάτι. Παρακολουθώ αυτά που λέτε και στην κρατηδιακή κυβέρνηση ε, υπηρέτησε ως Υπουργός Παιδείας και μάλιστα λειτουργήσα σε οικονομικά ε, δύσκολη εποχή. Ε, πάντοτε ζητούσαμε όταν υπάρχει κρίση όπως ε, και η οικονομική κρίση του 2009 σφίξαμε τα δόντια αλλά στο τέλος συμφωνήσαμε με περικοπές στον προϋπολογισμό ε, ανευπροηγουμένου η δυσκολία δεν είναι μόνο αυτή. Εγώ είδα συγκεκριμένα που περικόπτονται προγράμματα. Δεν είναι κακά προγράμματα αυτά που περικόπτονται, είναι εξαιρετικά και πήγαν και πολύ καλά. Ε, το COSMIS ε, είναι από τα καλύτερα προγράμματα για τις χώρες ε, που χρειάζονται για καινοτομία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κονδύλια. Κι όμως και αυτό περιεκόπη. Δεν έχω καταλάβει το γιατί, αλλά πάντως η περικοπή έγινε. Η αιτιολόγηση από το Συμβούλιο και πάλι η κριτική σας ήταν πολύ σωστή που εκφράστηκε και στον τριμερή διάλογο. Πολύ σωστά είπατε ότι όταν περικόπτονται προγράμματα θα πρέπει να είναι προγράμματα που σίγουρα δεν λειτουργούν. Αλλιώς θα πρέπει, όπως ήθιστε, να ε, ε, τροποποιούνται. Άμα ε, υπάρχει λόγος να συνεχιστούν και δεν έχουν πρόβλημα πρέπει να τροποποιούνται. υπήρχαν κάποια προγράμματα που ήταν προγράμματα βιτρίνα που δεν είχαν βιωσιμότητα και εμείς ασκήσαμε πίεση στην Κομισιόν για να βελτιώσει το πρόγραμμα. Και έγινε αυτό. Ε, πολλές φορές είχαμε επιτυχία. Τώρα βελτιώθηκαν προγράμματα και πάλι ε, προτείνονται περικοπές. Ε, αν ε, θέλει το Συμβούλιο να προετοιμαστεί με αυτόν τον τρόπο για το Brexit, εγώ είμαι κατά, γιατί αν γίνει άτακτο Brexit, τότε μπορεί να, βρίσκομαι, να βρισκόμαστε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βέβαια, αλλά να ζητάμε και να χρειάζονται τότε προγράμματα τα οποία ε, για τη Γεωργία για παράδειγμα να είναι τελείως διαφορετικά και πολύ μεγαλύτερα. Σίγουρα θα χρειαστεί μια συζήτηση για να δούμε τι θα κάνουμε τότε. Αλλά εκ των προτέρων να ακολουθούμε αυτή την πολιτική, αυτό είναι λάθος. Στο Άμυφ, για παράδειγμα, εδώ ε, έχουν ε, τελείως αλλάξει τα, τα κονδύλια. Δεν συμφωνώ σε προγράμματα όπου έχω 93% ε, ποσοστό απόρριψης ενώ ήταν εξαιρετικά προγράμματα και αιτήσει από όλη την Ευρώπη δεν μπορώ να δεχτώ την περικοπή σε αυτή την περίπτωση τα κράτη-μέλη οικονομικά είναι τώρα σε καλύτερη κατάσταση δηλαδή κανονικά θα έπρεπε να μπορούν να συμβάλλουν και σε τέτοια προγράμματα γι' αυτό πρέπει να συζητήσω με το Συμβούλιο ε, επί της ουσίας αυτών των ε, θεμάτων και προτάσεων. Αλλιώς ε, θα μας πούν ότι α, εσείς στο Κοινοβούλιο όλο θέλετε περισσότερα κονδύλια και συνολικά απορρίπτετε τις προτάσεις μας. Όχι, δεν θέλω να απορρίψω τις προτάσεις επειδή εγώ πάντοτε θέλω περισσότερα κονδύλια. Θέλω μια ωραία και συγκροτημένη αιτιολόγηση. Και θέλω συγκεκριμένα να επικρίνω το Συμβούλιο σχετικά με την ε, πρότασή του για τα προγράμματα. Και ε, θα συνεργαστούμε με τους συναδέλφους για να έχουμε καλά επιχειρήματα. Γιατί ε, η Φιλανδική Προεδρία μου το είπε ότι, σε ότι μα, εσείς θέλετε όλο, συνέχεια περισσότερα. Και ο Εμπλιάνο με βοήθησε εκεί και είπε και εσείς πάντοτε θέλετε λιγότερα. Ποτέ δεν έχει κάνει το Συμβούλιο μια πρόταση που να πει ναι, θέλουμε να επενδύσουμε σωστά. Δέκα χρόνια είμαι εδώ. Ποτέ δεν το έχω δει αυτό το πράγμα. Η επίκριση λοιπόν που μας κάνετε δεν μετράει ε, όταν πρόκειται για προγράμματα που δεν είναι καλά ή προγράμματα που δεν χρειάζονται. Θα συμφωνήσω με εκεί στην περικοπή. Αλλά για καλά προγράμματα, χρήσιμα προγράμματα, δεν μπορώ να δεχτώ την περικοπή. Θα πρέπει να υπάρχει πολύ σκληρή οικονομική χρηματοπιστωτική κρίση για να σφίξουμε τα δόντια και να πούμε ότι θα συμφωνήσουμε στις ε, ε περικοπές. Ευχαριστώ όμως πάρα πολύ για την ε, πάντα ε, υποστήριξη Και τώρα ο κύριος Πρέσα, ο οποίος είναι αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Προϋπολογισμών που βρίσκεται στην αίθουσα αλλά δεν με προσέχει αυτή την ώρα. Κύριε Πρέζα, καλώς ήλθατε. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτήν την ανταλλαγή απόψεων επί της εκθέσεως και της εισήγησης Χολμάγερ, που δείχνει ότι υπάρχουν θεμητές ανησυχίες για την πρόταση του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά το σχέδιο προπολογισμού 2020. Ο Επίτροπο Έτιγκερ συμμερίστηκε ορισμένε από αυτέ τι απόψει στο μέρη διάλογο τον Ιούλιο, οπότε συναντηθήκαμε και με το Συμβούλιο. Άρα, σε μεγάλο βαθμό, η Κομισιόν ευθυγραμμίζεται με τις θέσεις της εισηγήτριας, καθώς και των σκιωδών εισηγητών. Είναι πράγματι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς ε, τη λογική ε, περικοπών ε, σε στόχους που αποτελούν πολιτικές προτεραιότητες όπως είχαν αναγγείλει οι του Συμβουλίου. Άρα, από τώρα και μέχρι τη συνδιαλλαγή αργότερα υπάρχει κάποιο περιθώριο για να αντιστραφεί αυτή η κατάσταση που δεν συνάδει με τους πολιτικούς στόχους. Σε σχέση και με τον οικονομικό κύκλο πρέπει να τονίσουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος του ευρωπαϊκού προπολογισμού σε αντίθεση με τους εθνικούς προϋπολογισμούς είναι ε, προσανατολισμένο στις επενδύσεις. Ιδίως δε ε, σε περίπτωση οικονομικής ύφεσης που αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Άρα και αυτό είναι ένα επιχείρημα που κατατείνει προς την ενίσχυση του προϋπολογισμού και όχι στις περικοπές από πρακτικής πλευράς και διαδικαστικής πλευράς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα εκπονήσει την Επιτροπή Εκτελεστότητας, όπως το λέμε, το «Executive Letter, με τροπολογίες ε, δικές μας και του Κοινοβουλίου. Εμείς θα σχολιάσουμε την ε, δυνατότητα να εφαρμοστούν αυτές οι τροπολογίες και θα αναφέρουμε τις δυνητικές επιπτώσεις. Δηλαδή, μάλλον τις, θα δούμε ποιες είναι τροπολογίες του Συμβουλίου του Κοινοβουλίου. Και θα πάμε στη συνδιαλλαγή. Ο στόχος είναι βέβαια να έχουμε τους κατάλληλους πόρους που θα επαρκούν για την επίτευξη των πολιτικών στόχων. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Προσβλέπω σε καλή συνεργασία για τους επόμενους μήνες με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Thank you very much. I think uh, we Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι πράγματι ήταν ενδιαφέρουσα η συζήτηση, υπήρχε νομίζω συμφωνία ε, και τα συμπεράσματα λίγο πολύ κοινά. Σας ευχαριστώ λοιπόν για αυτή τη συζήτηση. Να πω ότι σε ό,τι αφορά τις δημοσιονομικές τροπολογίες στη θέση του Συμβουλίου πρέπει να έχουν κατατεθεί από τους ομονωμένους βουλευτές και από τις επιτροπές μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου. Οι ομάδες τώρα έχουν μία εβδομάδα παραπάνω στη διάθεσή τους. Η προθεσμία δηλαδή εκεί λίγη στις 12 Σεπτεμβρίου. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή Προπολογισμών θα διεξαχθεί εντός της εβδομάδας της 30 Σεπτεμβρίου. Κυρία Χολμάγερ, αν μου επιτρέπετε ε, ένα ερώτημα ή αν θέλετε να δώσω ε, έτσι μια κατεύθυνση στο τέλος. Είχαμε το δεύτερο γύρο των παραπρασκευαστικών δράσεων και των πιλωτικών προγραμμάτων. Ε, το πήραμε πίσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και δεν είμαι και τόσο ε, θετική. Γιατί αυτός ο δεύτερος γύρος ήταν πάρα πολύ σύντομος και Νομίζω ότι για όλα ήταν ε, αρνητικές ε, οι εκτιμήσεις και οι κριτικές, δηλαδή όλα τα απέρριψαν. Γι' αυτό ε, ζητώ από τους συναδέλφους που έχουν προσυπογράψει συγκεκριμένα προπαρασκευαστικές ενέργειες και πιλωτικά προγράμματα να έρθουν σε επαφή μαζί μου για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε Νομίζω ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν καταλαβαίνω. Ε, θέλει στο νέο ε, πι για την πολιτιστική κληρονομιά να τα έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα ε, και μιλάμε εδώ και για μια συγκεκριμένη πλατφόρμα και υποδομή σε θέματα τεχνολογίας πληροφοριών που θα πρέπει να θεσπιστεί. Και Πραγματικά δεν υπήρξε καλή κριτική. Ε, Τέλο πάντων, θα συζητήσουμε, μάλλον πρέπει να τα ξανασυζητήσουμε ε, και με τους συναδέλφους. Σίγουρα θα πρέπει να περιοριστούμε στα ουσιώδη, ε, να συμμαζέψουμε κάπως δηλαδή τις προτάσεις μα. και καλό είναι να εστιάσουμε στα βασικά ε, πού θα επιμείνουμε και πώς θα επιχειρηματολογήσουμε μετά. Αυτά πρέπει να τα ξαναδούμε. Ο πρόεδρο. Ευχαριστούμε κύριε Χολμάκη, οπότε θα τα πούμε ξανά στι 3 η ώρα. Και σα ευχαριστώ.